χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να μην ανταποκριθούμε θετικά στις προσδοκίες τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεών μας έχουμε μία αντιπροσωπεία από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας η οποία επισκέπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια της 21ης συνέντασης, συνάντησης των δύο κοινοβουλίων. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Τσαπεϊξίν, αντιπρόεδρο του Εθνικού Κοινοβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και ο κύριος ε, Ριβελίνη είναι οι δύο συμπρόεδροι μεταξύ των, ε, της συνάντησης των δύο αυτών κοινοβουλίων. Ο διάλογος αυτός συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή η νέα συνεδρίαση θα ενισχύσει τις διακοινοβουλευτικές μας σχέσεις έτσι ώστε να θίξουμε πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Εύχομαι οι δύο αντιπροσωπείες να μπορέσουν να συναντώνται συχνά έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε, να προσεγγίσουμε κοινά θέματα με κοινέ αποφάσεις. Ωρα. Εξ ονόματος της το λόγο έχει ο κύριος Σόλτς για δύο μισή λεπτά. Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπο και αντιπρόεδρε της Κομισιόν, συζητούμε στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο συχνά το θέμα της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ρωσία. Εξ ονόματος της δικής μου πολιτικής ομάδας, παρόλους τις επιφυλάξεις που είχαμε, ε, μπόρεσα να συμφωνήσω με το ψήφισμα που υποβάλαμε, από κοινού στο Κοινοβούλιο για τη διάσκεψη κορυφή. Θα ήθελα να σα πω ότι αυτή ήταν η πρώτη διάσκεψη κορυφή μετά την θέση ισχύ τη Συμφωνία τη Λισαβόνη και γι' αυτό ακριβώ η ρωσική πλευρά ελπίζει ότι θα υπάρχει μια πιο αποτελεσματική και αποφασιστική Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντί τη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε ο σημαντικότερο εταίρο τη Ρωσία. Το 2010 η Ρωσία σαν τελευταίο κράτη υπέγραψε την ε, Συμφωνία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ζητά την άρση των θεωρήσεων διαβατηρίων η Ρωσία. Εδώ και 7 χρόνια γίνουν διαπραγματεύσεις και δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αποτέλεσμα. Συμμερίζουμε απόλυτα την άποψη ότι με την πρόταση που υπέβαλε αυτή τη στιγμή η εταιρική σχέση για εξυγχρονισμό θα κινηθούμε προς μια στρατηγική συμφωνία εταιρική σχέσης. Αυτό όμως κατά γνώμη μου δεν αρκεί, ιδίω μια που το επίκεντρο των ευρωπαϊκών ε, μεταρρυθμίσεων Παραδείγματο χάρη δεν πρόκειται να προωθούνται οι προηγμένε ευρωπαϊκέ τεχνολογίε σε σχέδια στα οποία συμμετάχει και η κυβέρνηση της Ρωσίας. Εδώ δείχνουμε νομίζω ανεπαρκή ε, οραματικότητα και δεν ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να δούμε ότι η κύρια πρόκληση και από τις δύο πλευρές είναι το να ξεπεράσουμε την έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πολλά λόγια ακούγονται, δεν υπάρχουν όμως συγκεκριμένα και σοβαρά σχέδια που θα μπορέσουν να βοηθήσουν από όλες τις πλευρές την πολιτική, πολιτιστική ε, και οικονομική ζωή. Μία τελευταία παρατήρηση. Η ενέργεια και το περιβάλλον είναι κεντρικά σημεία για μία επικοδομητική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Συχνά αναφερόμαστε στην ενεργειακή πολιτική σαν ένα θετικό παράδειγμα τη δημιουργία εμπιστοσύνη, αλλά ακριβώ στον τομέα τη ενέργεια υπάρχουν πάρα πολλέ παρεξηγήσει και εδώ θα πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Έξω το ονόματο τη Ομάδα Ελευθερία και Δημοκρατία, ο κύριο Προβέρα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ρωσία είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε μια συμφωνία ε, εταιρικής οικονομικής συνεργασίας. Έτσι, θα μπορούσαμε να προωθήσουμε μια στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς. Ε, μιλώ για την ε, απελευθέρωση των θεωρήσεων, την, τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, τον έλεγχο του Ιράν, την ειρήνευση του Καυκάσου και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Πιστεύω ότι ο ενεργειακός μας τομέας δεν θα πρέπει να έχει θέματα ταμπού. Θα πρέπει να επιλύσουμε τον εφοδιασμό σε ενέργεια, γιατί αυτό θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία στο σχέδιο South Stream για τον ενεργειακό εφοδιασμό των επομένων ετών. Στις σχέσεις με αυτό τον σημαντικό οικονομικό εταίρο θα πρέπει να δράσουμε σε δύο διαφορετικούς τομείς. Καταρχήν να αντιμετωπίσουμε τα ιδεολογικά μας προηγούμενα και να δράσουμε με πραγματισμό ως προς τις διακρατικές σχέσεις. Εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων, ο κύριος Λεπέν για δυόμιση λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπο, σας συγχαίρω για τη νέα δυναμική που του, της νέας εταιρικής σχέσης η οποία υπογραμμίζει σε τι βαθμό είναι σημαντικός γεωπολιτικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ρωσία και χαιρετίζω τη συνεργασία με τη Ρωσία σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Κάποιες παρατηρήσεις θέλω να κάνω ωστόσο. Παρόλο που επαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλονται τα συμφέροντα και οι θέσεις των εταίρων τους υποτιμώνται ή αγνοούνται είτε πρόκειται για την ενέργεια ή για τον τρόπο ανάλυσης των συμπράξεων με την ε, από και την χώρες ε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στις ομιλίες τα περισσότερα, οι περισσότεροι εκπράσωποι των ε, ευρωπαϊκών κρατών καταδικάζουν μόνο τη Ρωσία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρησιμοποιούν πιο διπλωματική γλώσσα παρόλο, για την Κίνα, παρόλο που έχουμε και εκεί κατάφορες παραβάσεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εκτός από την Κίνα το ίδιο ισχύει και για άλλες χώρες. Σας θυμίζω το Αγκούστα Διά του Αγκούστα διότι έτσι πιστεύω ότι ε, κινείται σήμερα η Ρωσία εφόσον αποχώρησε ε, μπόρεσε να ξεφύγει το μαρξιστικό και το κομμουνιστικό καθεστώς παρόλες τις δυσκολίες και τα σημαντικές προκλήσεις που καλείται ακόμα να αντιμετωπίσει η χώρα αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να τη βοηθήσουμε να πετύχει τους στόχους της παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ασίας. Η χώρα ε, ε, πάρα πολύ, πάρα, πολύ συχνά ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη Ρωσία είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που ακολουθούσαμε στο παρελθόν. Και πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχουν προκύψει νέα ιστορικά γεγονότα μετά από την προοδευτική μετάφραση των ε, μυστικών αρχείων της Σοβιετικής Ένωσης, αρχεία που έχουν, ε, μας έχουν προσφέρει πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις σε πολλούς ανθρώπους σε ό,τι αφορά την περίοδο του ψυχρού πολέμου και μας δείχνουν ακριβώς ποιος υπήρξε ο ρόλος του κυρίου Γκορμπατσόφ με κίνδυνο να επαναλαμβάνω πράγματα που έχω ήδη πει, η Ρωσία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος για τις ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν οι σχέσεις μας. Η χώρα αυτή από πλευράς πολιτισμού και κουλτούρας, ιστορίας, γεωγραφίας, αμοιβαίων συμφερόντων, ε, κοινών κινδύνων ε, βρίσκεται πιο κοντά από εμά σε σχέση με πολλές άλλες χώρες που σπρώχνεται να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουμε τώρα το λόγο στους άλλους ομιλητές και θα ήθελα να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας γιατί έχουμε καθυστερήσει. Για δύο λεπτά έχει το λόγο κυρία Όμεν Ρόιτον. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν για να φτάσουμε σε μία σαφή πρόταση ψηφίσματος όπως την παρούσα. Κυρία Αντιπρόεδρε, στο ψήφισμα αυτό επικρίνουμε ορισμένες πτυχές της συνάντηση στο Ροστόφ. Δηλαδή είχαμε πενιχρά αποτελέσματα. Και αυτό είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο, διότι η Ρωσία προτιμά διμερείς συμφωνίες με τα μεμονωμένα κράτη παρά μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλά με ενία φωνή. έδρασε ενιαία πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε λόγος για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης, οικονομικής εταιρικής σχέσης. Αυτό που έχει σημασία είναι να εξεύρουμε μια δεσμευτική, ένα δεσμευτικό τρόπο συμφωνίας πέρα και μαζί με το ενεργειακό. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης σεβασμός και τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως προς τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης είναι ύψης της σημασίας και για εμάς και για τους ε, ε, Ρώσους. Μιλήσαμε για εξυγχρονισμό. Εγώ θεωρώ ότι αποκλειστήκαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα προγράμματα εξυγχρονισμού δεν είναι απόλυτα σαφή. Βεβαίως ε, προετοιμάζονται πρωτοβουλίες γιατί για τον εξυγχρονισμό της ρωσικής οικονομίας θα πρέπει να υπάρξει, να γίνει πρωτίστως μία ε, συμφωνία στον ενεργειακό τομέα και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ως προς τον κοινό οικονομικό χώρο, το πρόγραμμα εξυγχρονισμού δεν ε, είναι ίδιο με αυτό που συμφωνήθηκε στους τέσσερους κοινούς χώρους. Εν πάση περιπτώσει, στο ψήφισμα θα πρέπει να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το έχουμε υπενθυμίσει πολλές φορές και υπάρχουν και τροπολογίες επί του θέματος που θα ήταν σκόπιμο να υπερψηφιστούν. Λυπάμαι, λέει η Πρόεδρος, αλλά θα πρέπει να σας διακόπτω, διότι δεν μπορείτε να υπερβαίνετε το χρόνο σας περισσότερο από 40 δευτερόλεπτα. Ο κύριος βόποτα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπα, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που μας κάνατε εδώ. Με παρουσία πολύ ανοιχτή και σαφή. Ε, κατεδείξατε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία θα ήθελα να μπορούσαμε να έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση. Θα ήθελα να σας πω όμως ταυτόχρονα ότι η Ρωσία είναι ένας εταίρος που δυστυχώς δεν τηρεί πάντα όλες τις συμφωνίες. όσον αφορά τη Γεωργία. Και ακριβώ κάποιο που ήταν πάρα πολύ επικριτικό όσον αφορά τι δραστηριότητε τη Γεωργία στο τελευταίο πόλεμο, ομολογώ ότι λυπούμε που η Ρωσία τώρα δεν τηρεί τη συμφωνία με τη Γεωργία γιατί αυτό βέβαια αποδυναμώνει τη θέση της Ρωσίας και τη δυνατότητα της Ρωσίας να δρά ειρηνοποιά στον χώρο αυτό. Τώρα η κατάσταση που έχουν στο Κυρκιστάν είναι κρίσιμη και θα ήταν ίσως ε, αρμόζων προς τη Ρωσία να βοηθήσει να επιληθεί το πρόβλημα. Ε, όσον αφορά το θέμα και σε σχέση με την ΟΗΕ θα πρέπει να πούμε στη Ρωσία ότι εμεί θέλουμε την εταιρική σχέση μαζί τους αλλά η Ρωσία θα πρέπει να τηρεί και τους κοινούς κανόνες που έχουμε αναπτύξει με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών και να τηρεί τις συμφωνίες που έχουν συμφωνηθεί με τη Σοβιετική Ένωση. Θα ήταν καλό να αναπτυχθούν διαφορετικά οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βλάψουμε τις σχέσεις Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αναπτύσσονται θετικά συνεχώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Λάμστορφ. Κυρία Αντιπρόεδρε, αυτά που είπε ο συνάδελφος Σβόβοντα είναι και η στάση της δικής μας ομάδας. Εμείς θέλουμε μια σταδιακή εταιρική σχέση με τη Ρωσία, από την άλλη μεριά πιστεύουμε δεν την έχουμε. Γιατί βάσει των αξιών που δεν συμμεριζόμαστε με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να καταλήξουμε στρατηγική ε, εταιρική σχέση. Υπάρχουν όμως ευκαιρίες και ευκαιρίες που είναι στη δική σας θητεία Βαρόνια, που δεν έχει ίσως προκατοχό σα. Γιατί αυτό που έχουμε στη Ρωσία είναι μια δυτική πολιτική εντό εισαγωγικών που είναι πιο επιδομητική αυτό που βλέπαμε στο παρελθόν. Παραδείγματο χάρη των προβλημάτων στα σύνορα με την Ορβηγία στην Αρκτική η συμφωνία με την Ουκρανία όσον αφορά τις ε, βάσεις της Σεβαστούπολη. Μια συμφωνία που ελπίζουμε να σταθεροποιήσει την ε, τροφοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από τη Σοβιετική Ένωση, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο και επίσης τη συμφιλίωση της Ρωσίας με την ε, Πολωνία, παραδείγματο χάρη η κρατική τηλεόραση στη Ρωσία έδειξε δύο φορές την ταινία Κατίνε και αυτό είναι πάρα πολύ επιδοφόρο. Φαίνεται ότι πια η Ρωσία αναγνώρισε ότι τα κύρια της ε, προβλήματα βρίσκονται στο Νότο και στα Ανατολά. Αναφέρθηκε το Ιράν ήδη και θα πρέπει ίσως να δούμε τι θα γίνει σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν ε, τι θα γίνει με μια νέα ε, κρατική συμφωνία. Υπάρχουν ελπίδες και ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερες σχέσεις και θα προχωρήσουμε πιο μια στρατηγική ε, εταιρική σχέση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Χατάλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης και όλη την ομάδα που ταξίδευσε στη Ρωσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που διαπιστώνω ότι το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής μας συζήτησης. Έχουμε ωστόσο κάποιες ανησυχίες σχετικά με το ψήφισμα που θα ψηφιστεί αύριο. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να ρυθμιστούν. Έχουμε πολλές επαφές μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου και αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε άτομα αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη περίπτωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους Ρώσους συναδέλφους. Αναφέρθηκε σε δύο περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν παράδειγμα ατόμων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα με κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Ρόστοφ που έγινε αυτή η σύνοδος κορυφής δεν επιτράπησαν οι διαδηλώσεις ε, των πολιτών οι οποίοι όμως ήθελαν να ε, προασπίσουν το άρθρο 31 του ε, Ρωσικού Συντάγματος. Ευχαριστώ κυρία Ούτελα. Ο κύριος Κούρσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εάν δεν υπάρξει συγχρονισμός της Ρωσίας με την χρήση των νέων τεχνολογιών δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο ύψος του ε, μεσοόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται ωστόσο αυτό διότι το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής καθόλου δεν είναι ικανοποιητικό και νομίζω ότι θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση έως ότου τηρήσει πιο σκληρή στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζοντας και προβάλλοντας ορισμένες σημαντικές αξίες. Γι' αυτό η νέα εταιρική σχέση με τη Ρωσία πρέπει να συμπεριλάβει κάποιες ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να λέει σαφώς ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστεί μαζί μας η Ρωσία εάν βελτιώσει τη στάση της σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί δεν αντιδράσαμε στις διαδηλώσεις στην Αγία Πετρούπολη ή στη Μόσχα δεν αρκεί να λέμε, να λέμε ωραία λόγια. Πρέπει τα λόγια αυτά να συνοδεύονται με συγκεκριμένες πράξεις. Ο κύριος Μπέλντερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Από την εποχή του, του Πέτρου του Μεγάλου η Ρωσία προσπαθεί να προβάλλει έναν εξυγχρονισμό για τη χώρα. Και αυτό διαφαίνεται σε όλη της ε, την πορεία. Φάνηκε και με την τελευταία συνάντησή μας στο Ρόστοφ Οντών. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη το ότι θα πρέπει να πείσουμε τους επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας για την ε, σημασία του εξυγχρονισμού, η οποία θα πρέπει να είναι αμφίδρομη, αλλά αυτό όχι μόνο μέσα στα πλαίσια των υλικών αγαθών, αλλά και των αήλων, δηλαδή με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαφορετικά θα βρεθούμε σε λάθος δρόμο, κάτι το οποίο θα έχει ολέθριες συνέπειες. Νομίζω ότι το μοντέλο Πούτιν δημιουργεί τριβές και στις σχέσεις με την Ουκρανία. Λίζεκ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ε, λέει Διάστον, είναι καλό το ότι συζητούμε με τη Ρωσία. Χρειάζεται ο διάλογος με τη Ρωσία και όλοι οι συνετοί άνθρωποι θα συμφωνήσουν με αυτό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει αυτό το διάλογο με τη Ρωσία. Η Ρωσία αλλάζει, το ελπίζουμε τουλάχιστον. Και ελπίζουμε ότι όπως είπε ο κύριος Μετβέντεφ ότι θα υπάρξει η δικτατορία του κράτους δικαίου και ότι οι επιχειρηματίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνουν επενδύσεις ή εμπόριο με την ε, Ρωσία θα ξέρουν ότι ε, το νομικό καθεστώς θα στηρίζει και δεν θα παρεμποδίζει τη δραστηριότητά τους. Μέχρι σήμερα υπήρξαν πάρα πολλά νομικά θέματα, νομικά προβλήματα στη Ρωσία. Όταν μιλάμε με τη Ρωσία πρέπει να το, το, το υπενθυμίζουμε αυτό στους Ρώσους. Χαιρόμαστε που συνεργάζεται η Ρωσία με τα ευρωπαϊκά κράτη, με τον ΝΑΤΟ, τον Ηνωμένα Έθνη, τον, την, τις Ηνωμένες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή για θέματα παγκόσμιας ασφάλειας. Αλλά μας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί ή ληφθεί υπόψη όλα τα προβλήματα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τι γειτονικέ χώρες. Μας απασχολεί το γεγονός ότι υπάρχουν Ρώσοι πολιτικοί οι οποίοι θέλουν να αποκαταστήσουν την ε, ρωσική αυτοκρατορία. Ε, στην περίπτωση της Γεωργίας ε, ειδικότερα και πρέπει λοιπόν να παρεύουμε και να του υπενθυμίσουμε ότι αυτά δεν είναι πράγματα που επιτρέπονται πλέον σήμερα. Frau Präsidentin, Lady Ashton. Κύριε Πρόεδρε, Λέδη Άσον, αγαπητοί συνάδελφοι, η διάσκεψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία ε, οδήγησε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ιδίω όσον αφορά τη συγκεκριποίηση τη ε, εταιρική σχέση εξυγχρονισμού. Και χαίρομαι που ο διάλογο ε, μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών θεωρείται μία από τι προτεραιότητε μέσα στα πλαίσια τη εταιρική σχέση αυτή για τον εξορισμό. Θα μέλο τη αντιπροσωπεία με την Ρωσία ηγήθηκα μια συνάντηση στο ΠΕΝ πρόσφατα που ασχολήθηκε ακριβώς με αυτό το θέμα και για άλλη μια φορά είδαμε η πρόοδος έχει επιτελεστεί τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία αλλά πόσα πρέπει ακόμα να γίνουν και πόσα θα πρέπει εμείς βάσει των εμπειριών μας καλών ή και όχι τόσο καλών μπορούμε να συμβάλλουμε. Ανταλλαγή απόψεων είναι πάρα πολύ σημαντική για μας Κεντρική σημασία. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μια εταιρική σχέση χωρί την ανταλλαγή ανθρώπων και γι' αυτό λυπήθηκα που δεν προχώρησε περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τι θεωρίε των διαφατηριών. Θα πρέπει τώρα να ορίσουμε συγκεκριμένου στόχου για του οποίου θα πρέπει να συνεργαστούν από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία. Το πρόβλημα δεν είναι να τηρήσουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα ή κάποια σειρά προτεραιότητος, αλλά θα πρέπει να είμαστε στη δυνατότητα να ορίσουμε ακριβώς τα κριτήρια ο καθένας δηλαδή στη Ρωσία να μπορεί να ξέρει αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, αν επιληθούν τα συγκεκριμένα προβλήματα θα υπάρχει απελευθέρωση από τις ορίσεις διαβατηρίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαρνέτσκι, για ένα λεπτό relacje unii z to musi być μας πρέπει να είναι φίδρομες. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της χώρας, αλλά πρέπει και εκείνοι να μας δώσουν κάτι σε αντάλλαγμα, να βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα για τους επενδυτές μας και να υπάρξει κάποια νομική βεβαιότητα και σταθερότητα. Λυπάμαι ότι στη διάρκεια αυτής της Συνόδου Κορυφής επικράτησε ένας μονόδρομος. Δώσαμε εμείς πράγματα χωρίς να πάρουμε τίποτε σε αντάλλαγμα. Σε αυτό το κοινό ψήφισμα υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας. Δεν, αναφέρεται, δεν αναφέρονται πουθενά συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αναφερθούν τα ονόματα, θα πρέπει να ε, δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα που είναι πολλά. Εάν η Άγγελα Μέρκελ και ο πρόεδρος Μεντιβέντεφ συμφωνήσουν ε, για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας θα πρέπει όλοι να μιλάμε με μια ενιαία φωνή. Μίλαν μόνο e για 1,5 λεπτό. Σας παρακαλώ συνάδελφοι να ησυχάσετε λίγο. Η σημασία των σχέσεων μας είναι αυταπόδεικτη σε όλους τους τομείς οικονομικό, ενεργειακό και ούτω καθεξής, αν λάβουμε υπόψη ότι η Ρωσία είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της αντιπυραυλικής ασπίδας που προβάλλει η Ρωσία. Σε αυτά τα πλαίσια μιλάμε και για τη στάση της Ρωσίας ως προς το Ιράν, όπως διαφάνηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας και το τελευταίο του ψήφισμα. Λυπάμαι κυρία Άστον, διότι δεν επιτεύχθηκε μεγαλύτερη συμφωνία με τη Ρωσία, γιατί μιλάμε για την ενδεχόμενη προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, κάτι το οποίο δεν διασαφηνίστηκε. Θα πρέπει να επιλύσουμε τις ε, ενεργειακές σχέσεις και το εμπόριο, τις σχέσεις ενεργειακού κυρίως εφοδιασμού. Θα πρέπει να δεχτούμε τον εξυγχρονισμό της Ρωσίας, αλλά εταιρική σχέση σημαίνει ότι υπάρχει αμφίδρομος χαρακτήρας. Κάτι το οποίο δεν ισχύει Χαίρομαι διότι η Προεδρία συμπεριλαμβάνει και την συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω τα νέα μέσα της συνθήκης της Λισαβόνας να μας επιτρέψουν κάτι τέτοιο έτσι ώστε να προωθήσουμε μια πραγματικά ενιαία πολιτική και να μιλάει η Ευρώπη με μια φωνή έναντι όλων των εταίρων. Συνάδελφοι, βρισκόμαστε στη λήξη της συζήτησης. Θα ήθελα σας παρακαλώ να ησυχάσετε, να, είσαστε, να προσέρχεστε με ησυχία στην αίθουσα. Ο κύριος Βιτζένιν για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθείτε να βάλετε τάξη στο ενέθουσα, αλλά φοβάμαι ότι ο θόρυβος διαρκώς θα αυξάνεται. Κυρία, είπατε εκπρόσωπο. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε για την συνάντηση με τη Ρωσία μια συνάντηση που μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα που υπήρξε επικοδομητική με λιγότερη ένταση, περισσότερο ρεαλισμό και περισσότερο σεβασμό και από τις δύο πλευρές. Αυτό το νέο κλίμα θα οπωσδήποτε θα ενισχύσει, θα βελτιώσει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Υπάρχει οπωσδήποτε κάποια διάσταση απόψεων ως προς τις αρχές τις οποίες πρεσβεύουμε η ΜΕΝ και η ΔΕΑ, αλλά παράλληλα έχουν τεθεί περισσότεροι στόχοι που επιδιώκουμε από κοινού. Υπάρχει ένα ευρύτερο φάσμα που μπορούμε να αναλάβουμε από κοινού. Δεν συμφωνώ με του συναδέλφου ότι το ψήφισμα που πρόκειται να ψηφίσουμε είναι αδύναμο. Όχι, είναι ένα καλό ψήφισμα, κάτι το οποίο έχουμε καιρό να δούμε και πιστεύω ότι αυτό το ψήφισμα δείχνει, παρουσιάζει με ουσιαστικό τρόπο τα αποτελέσματα αυτή τη Συνόδου Κορυφή. Η εταιρική σχέση, για την εταιρική σχέση είναι σημαντική η πιο στενή επικοινωνία με τη Ρωσία που θα μας επιτρέψει να λύσουμε ε, προβλήματα που εκκρεμούν για πολύ καιρό σε σχέση με τις διάφορες χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την εταιρική σχέση. Ως προς το Catch the Eye θα δώσουμε το λόγο μόνο σε έναν ομιλητή από κάθε πολιτική ομάδα διότι έχουμε καθυστερήσει πολύ. Αρχίζουμε με τον κύριο Βαϊντέρε για ένα λεπτό. sadarbība Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συνεργασία με τη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Η νέα συμφωνία για την εταιρική σχέση πρέπει να είναι νομοθετικά νοσβευτική και πιο συγκεκριμένη. Η συνεργασία για τον εξυγχρονισμό πρέπει να είναι διμερής και ισόρροπη και αναλογική και ω μέλο τη Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να υπογραμμίσω στα 115, σε 115 δικαστικέ αποφάσει κατά τη Ρωσία του Διεθνού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η ε, Ρωσία παραδέχθηκε με την ανοχή της αλλά δεν καταβλήθηκαν καθόλου αποζημιώσεις για περιπτώσεις ε, για ορισμένες περιπτώσεις που άνθρωποι πέθαναν ε, στη φωτιά στη Λετωνία μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα η ρωσική κυβέρνηση αναγνώρισε την πράξη της αλλά δεν καταβλήθηκε καμία αποζημίωση. Έχουμε λοιπόν μια τελείως διαφορετική άποψη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάσκου για ένα λεπτό. To my mind, in terms of... Uh, Κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά τα αποτελέσματα της διαπιπτώσεως, η διάσκεψη κορυφής ε, γερμανο-ρωσική ε, κορυφή θα ήταν πιο αποτελεσματική ίσως από εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί τα θέματα ασφάλειας θα πρέπει να συζητιούνται πιο μόνιμα μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας και της ΕΕ εφόσον οι, και τα δύο μέρη εννοούν τα ίδια πράγματα όταν ζητάνε αυτά τα θέματα θα πρέπει να έχουν ανταλλαγή απόψεων επίσης για διεθνή τρέχοντα προβλήματα. Εγώ μια που είμαι καθηγητής ε, εξωτερικής πολιτικής έχω να σας πω ότι δεν μπορώ ποτέ να ξεχνάω ότι οι λεπτομέρειες που είναι τα πιο δύσκολα τα έχετε αφήσει στα κατώτερα στρώματα της διαπραγματευτικής ομάδας. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Μότσερ για ένα λεπτό. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πολλά δεν πέτυχε η διάσκεψη κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία. Η συμφωνία αυτή για την εταιρική σχέση εξυγχρονισμού υπάρχει μόνο επί χάρτου και δεν ξέρει κανένα πού θα βασιστεί. Εκτός αυτού δεν αναφέρεται κανένα χρονοδιάγραμμα και κανένα συγκεκριμένο σχέδιο. Όπως ξέρουμε όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό οι σχέσεις με τη Ρωσία να εμβαθυνθούν γιατί ιδίω όσον αφορά τι ενεργειακέ σκέψει, η Ρωσία είναι πιο σημαντικό εταίρο τη Ευρώπη. Ε, εάν καταβάλουν προσπάθειες για να δεσμευτεί η Ρωσία προς τις άλλες εταιρικέ ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου φαίνεται θα ήταν αντιπαραγωγικό. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις ανάγκες για κάθε χώρα για να δούμε και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ήδη το 2004 δεν ήταν και τόσο επιτυχές. Το να συζητιέται τώρα η Γάζα, το Ιράν και η μείωση των ε, πυρήνων ε, κρίσης με κάνει να ρωτιόμαι γιατί δεν συζητήθηκε το θέμα του Κυργιστάν όπου εκεί καταραίουν οι κρατικές δομές. Ευχαριστώ. Διακόπτη πρόεδρος. Κλείνει η διαδικασία των παρεμβάσεων ενός λεπτού και δίνουμε το λόγο στην Αντιπρόεδρο Άστον και τη ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη για την φασαρία που επικρατεί στην αίθουσα. Σας παρακαλώ συνάδελφοι, λίγη ησυχία. Έχετε το λόγο. Thank you, Madam President. I hope... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you, Madam President. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω ότι όποιος θέλει να ακούσει τα συμπεράσματα για τη συζήτηση να μπορεί να το κάνει. Εγώ θα συγκεντρώσω την προσοχή μου σε ορισμένα βασικά θέματα που έθεξε μια σειρά βουλευτών. Καταρχήν τη σχέση μεταξύ της ε, εταιρικής συμφωνίας εξορισμού και της ε, συμφωνίας ε, πολιτικής συνεργασίας δεν είναι ε, μεν το ένα σε θέση να αποκλείσει το άλλο, αλλά εγώ θέλω να υπάρχει σημαντική προοδό όσον αφορά ιδίω τα οικονομικά και εμπορικά κεφάλαια. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία μαζί με την απαρχή της εταιρική σχέσης για τον εξυγχρονισμό. Μια απαρχή κάναμε, τίποτα άλλο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, το είπε ο κ. Σεβερή νομίζω. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό. Κύριε Κόσκερη, συμπεριλαμβάνονται τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν αναφερόμαστε μόνο στα τεχνικά πλεονεκτήματα που θα θέλει να αποκτήσει η Ρωσία. Είναι πολύ πιο ευρύ όσον αφορά μεταρρυθμίσει στο δικαστικό. Και επίσης θα ήθελα να σας ε, αναφέρω στην ε, τελική δήλωση για τη διάσκεψη κορυφής. Εκεί νομίζω συμπεριλαμβάνονται αυτές οι ιδέες και κύριε Μπέλτερ μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε άμα διαβάσετε συμπεράσματα. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε με μια φωνή όπως ιδίως ανέφερε η κυρία Ουμεν Ρόιτν. Είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να διαβλέπουμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και με συνέπεια σε διάφορους τομείς και νομίζω ότι η Ρωσία προτιμά να μπορεί να μιλά με το σύνολο των 27 χωρίς αυτό να αποκλίνει από τις σχέσεις που έχει με ορισμένες χώρες διμερώς, αλλά είναι πολύ πιο δυνατό να επιδράσουν μέσω της συνομιλίας με τους 27, ιδίως για οικονομικά θέματα, παρά αν είχαν επικοινωνία μόνο με μεμονωμένα κράτη. Όπως είπε ο κ. κ. Λεπέν και ο κ. Μάναμεν, ε, έχω να πω ότι όταν συζητάμε παραδείγματο χάρη με τον Λάβρο για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε πιο στενά για θέματα ε, ανά τον κόσμο το θέμα του Ουσβετικιστάν και του Κυριστάν τώρα μόλις παρουσιάστηκε στις τελευταίες 48 ώρες δεν ήταν τότε επίκαιρο εμείς όμως εξακολουθούμε να έχουμε επικοινωνία με τη Ρωσία εγώ έμεινα σε επικοινωνία τηλεφωνικά και για το Καζακστάν και με άλλες χώρες ο κύριος Στάνη και ο κύριος τα ιδιαίτερα αναφερθήκαν στην Ουκρανία. Χθε συνάντησα τον Ουκρανό Πρωθυπουργό, ιδίω για να συζητήσουμε τρόπου με του οποίου θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία. Κατανοώ ότι η Ουκρανία είναι ένα σημαντικό βήμα για μα και για το τι κάνουμε σχετικά με τι θεωρήσει στην ε, περιφερειακή. Για στην αρχή είτε συζήτησε ο κ. Μπροκ είπε ότι πραγματικά εργαζόμαστε με συνέπεια με όλους τους εταίρους μας της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης, ούτως ώστε να μην δημιουργήσουμε απαράδεκτες ανισορροπίες. Κύριε ε, Φλέκενστάιν, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και η κίνηση της Ρωσίας προς την ΠΟΕ, όπου θα πρέπει να ξαναεξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθούν στην ε, ΠΟΕ. Τώρα, κατά πόσον θα έχουν μια εταιρική σχέση με το Καζαστάν και θα, από κοινού θα ενταχθούν εκεί, δεν ξέρω. Ο κ. Σύμβουλο θα μα βοηθήσει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Εκτό αυτού, τελειώνοντα, το η γεωργία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ. Και αποδίδω φόρο τιμή στο πιο για αυτό που είπε. Τέλος πρόεδρε, η ενέργεια είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο θα πρέπει να παραμείνουμε σε στενή ενεστερική σχέση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε. Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος. Με τη λήξη της συζήτησης η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες.